Καθίστε παρακαλώ. Ich Επανάληψη της Συνόδου της 7ης ε, Ιουλίου. Αξιότιμοι συνάδελφοι στις 24 ε, Αυγούστου στη μέση της Ιταλίας. Η Ιταλία μάλλον επλήχθη από έναν ισχυρό σεισμό και Σημειώθηκαν ζημιές σε 70 και παραπάνω χωριά. Κάποιες κοινότητες καταστράφηκαν ολοσχερός μάλιστα. και είδαμε με φρίκη τις εικόνες από την Αματρίτσε, Πασκάρα, Τρόντο και πάνω από 3.000 άτομα μέσα σε μια νύχτα βρέθηκαν χωρίς ε, κεραμίδι πάνω το κεφάλι τους και βρέθηκαν ε, μπροστά στα συντρίμια της ζωή τους. Εξ ονόματο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα ήθελα καταρχάς να τιμήσω τις ε, υπηρεσίε έκτακτη ανάγκη, την πρεσβεστική, τις ιατρικέ υπηρεσίε, τους εθελοντές, να σας ευχαριστήσω όλους τους. Όλους εκείνους που δεν δίστασαν να κάνουν τα πάντα για να δώσουν τις πρώτες βοήθειες και να προστατεύσουν αυτούς που επλήχθησαν η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα σταθεί στο πλευρό των ανθρώπων αυτών με πλήρη ελληνική. Ο σεισμός ε, προκάλεσε ισχυρές ε, ηλικές, μεγάλες ε, ηλικές ζημιές. Χωριά ισοπεδώθηκαν και δεν είναι μόνο αυτά τα χωριά, ξέρετε, η Ιταλική πολιτιστική κληρονομιά, αλλά και η Ευρωπαϊκή πολιτισμική κληρονομιά. Αλλά ξέρετε, οι υλικέ ζημιέ καλύπτονται. Αυτό που μένει είναι ο ανθρώπινο πόνο, ο πόνο των οικογενειών, των 300 περίπου, 300 περίπου θυμάτων. Τα χωριά μπορούν να ανοικοδομηθούν και σίγουρα θα ανοικοδομηθούν. Αλλά το κενό που αφήνουν πίσω τους οι νεκροί δεν μπορεί να γεμίσει. Η αλληλεγγύη λοιπόν με τον συνάνθρωπό μας και η αλληλεγγύη για τον Ιταλικό λαό θα με οδηγήσει να σας ζητήσω σε, να σηκωθείτε σε, για ένα λεπτού σιγή. danke Σας ευχαριστώ. Τα πρακτικά λοιπόν της 7 η Ιουλίου είναι στη διάθεσή σα Δεν ξέρω κατά αυτόν. Έχουν εκριθεί λοιπόν τα πρακτικά. Κυρίες και κύριοι, θα θυμάστε ότι στις 6 Ιουλίου ε, κατά του κ. Κόρβιν Μίκε επιβλήθηκαν κύριο